η ισότητα ανδρών και γυναικών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν προκαταλήψεις ανάμεσα στα δύο φύλλα που, και μισογυνισμός. Θα πρέπει να σταματήσει επίσης η λεκτική βία, αλλά και η φυσική βία. Και οι άντρε θα πρέπει να πολεμήσουν για την ισότητα. Είναι υποχρέωσή μας. Η στρατηγική που προτείνεται θα έχει τεράστια αξία και θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε χάρη σε αυτήν όλοι μας. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριο Κράχ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ο μεγάλος Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλ Ρέγαν είπε μία φορά ότι οι δέκα χειρότερες λέξεις στα αγγλικά είναι ε, ε, «Γεια σας, είμαι από την κυβέρνηση και ήρθα να σας βοηθήσω». Το θέμα το, της των σχέσεων των φίλων είναι από τις πιο ιδιωτικές ε, ε, λεπτές σχέσεις των ανθρώπων. Η σκέψη ότι θέλει η Κομισιόν να παρέμβει μια στρατηγική είναι ανεξάρτητο από το αν η στρατηγική είναι σωστή ή όχι, αν λέει σωστά πράγματα. Είναι λάθος η παρέμβαση του κράτους στην ιδιωτική σφαίρα είναι αντιφιλελεύθερο, είναι ολοκληρωτική προσέγγιση. Οι συνάδελφοι της αριστεράς ξεκαθάρισαν ότι εδώ πρόκειται για ε, ένα σχέδιο που έχουν ε, προς την καταστροφή, υπέρ της καταστροφής της ε, οικογένειας και της προώθησης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Και ακριβώς εδώ είμαστε αντίθετοι. Ευχαριστώ πολύ ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Πέτερ Χάνσεν ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω να ε, είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για το σχέδιο. Χάρηκα που το υποβάλατε. Ελπίζω αυτή η στρατηγική να μην δώσει κενά μηνύματα στις γυναίκες, να δείξουμε ότι τις παίρνουμε στα σοβαρά. Ήρθε η ώρα γι' αυτό. Είναι σημαντικό να φτάσει το μήνυμα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, να περάσει το μήνυμα ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση ε, στο ε, στη Δεν ε, καλύπτονται όλες οι γυναίκες από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης πάρα πολλές πληρώνονται λιγότερα από τους άνδρες συναδέλφους. Η στρατηγική της Κομισιόν είναι το πρώτο βήμα και το δεύτερο βήμα είναι συγκεκριμένη νομοθεσία για να αλλάξει η κατάσταση. Μην ε, φοβηθούμε τις κυρώσεις γιατί είναι σαφές ότι χρειάζονται. Χρειάζεται δράση υπέρ των Ευρωπαίων γυναικών. Περιμένω τα επόμενά σας βήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η ισότητα των φίλων είναι θέμα δικαιοσύνη για τι γυναίκε. Ακόμα και στι πιο συντηρητικέ κοινωνίε βλέπουμε θεραλέ γυναίκε να θέτουν το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών στο τραπέζι αλλά δεν εισακούνται πάντοτε τα αιτήματά τους. Οι πολιτικοί δίνουν μεγαλοσχήμονες υποσχέσεις, αλλά τελικά δεν αναγνωρίζουν επαρκώς το ρόλο των γυναικών στην ε, κοινωνία και την οικονομία. Αν δεν πετύχουμε τους, στρατηγικούς, ε, τους στόχους στρατηγικής για τις γυναίκες, θα αποτύχουμε έναν του μισού πληθυσμού θα πρέπει να βασιστούμε σε ένα αυθεντικό διάλογο με τους ε, πολίτες, άρα να εισακούσουμε τις γυναίκες σε σχέση με τη μελλοντική τους προοπτική. Θα πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη με γυναίκες που μάχονται για την ισότητα στο πλαίσιο των δικών τους κοινωνιών. Η στρατηγική της Κομισιόν είναι μια καλή αφετηρία ε, για ανάληψη δράσης και είναι και μια, ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ο φορέας εκείνος ο οποίος θα δημιουργήσει ε, ελπίδα για τις γυναίκες. Η... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είχα προετοιμάσει ένα ε, μια ομιλία σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι εδώ είναι, οι περισσότερε ομιλήτρες είναι, είναι γυναίκες και σκέφτομαι ότι κάθε φορά που μιλάμε σε αυτό το σώμα για χρήματα ε, οι πυράβλους ε, το, το λόγο έχουν κυρίως οι άνδρες. Ενώ όταν μιλάμε για ισότητα των φίλων, ομιλήτριε είναι κυρίως οι γυναίκες. Τώρα, το θέμα των διακρίσεων και της βίας αφορά τους άνδρες. Η... Πρόκειται για... το πώς ε, οι κόρες μας ε, πέφτουν θύματα βίας, οι γυναίκες μας ε, κερδίζουν λιγότερα χρήμα από τους άντρες τους, οι γιαγιάδες μας οι οποίες έχουν χαμηλότερες συντάξεις γιατί όλη τη ζωή κέρδισαν λιγότερα χρήματα από τους άνδρες συναδέλφους τους. Άρα, συνάδελφοι, σας απευθύνω μια έκκληση. Ας δείξουμε αλληλεγγύη έναντι των γυναικών που μάχονται για τα δικαιώματά τους, γιατί αυτό θα επηρεάσει όλες τις γυναίκες που γνωρίζουμε εμείς προσωπικά. Θέλετε να δεχτείτε την μπλε κάρτα, ε, το ερώτημα... Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ε, δηλώσεις. Μια προσωπική ερώτηση. Τι νομίζετε ότι μπορεί να κάνουν οι άνδρες για να εθαρρύνουν τις γυναίκες. Θεωρείτε ότι οι άντρες θα πρέπει να ε, πάνε στην άκρη προκειμένου να προβληθούν οι γυναίκες. Ποια είναι η προσωπική σας θέση. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς προκειμένου να ενισχύσετε την θέση των γυναικών ως πολιτικός και εντός της ε, πολιτικής σας ομάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δοθεί απάντηση από τον κύριο Πέτρα. Θα πρέπει να στραφούμε προς τα πίσω, να δούμε ότι κάθε μέρα άντρες και γυναίκες μένουν στο περιθώριο. Εμείς ως πολιτικοί έχουμε ευθύνη για αυτούς τους ξεχασμένους. Ε, εμείς ως άρενες πολιτικοί έχουμε επιπλέον εξουσία. Πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες, να τις απελευθερώσουμε, να τις καταστήσουμε ίσες. Τίποτα άλλο. Όχι οι ανώτερες ή κατώτερες ίσες. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Και τώρα ο κύριος Σιμέτσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Είμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση. Από τη μία βλέπουμε την αυξανόμενη πίεση του κοινού για την ανισότητα των φύλων και απ' την άλλη, σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε μια ανησυχητική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά όταν βλέπουμε τα νούμερα και του οικονομικού δείκτε. Σχεδόν σε κάθε οικονομικό δείκτη οι γυναίκε τα πάνε χειρότερα. Έχουν χαμηλότερου μισθού κατά 16%. Έχουν ε, δύο φορές λιγότερη εκπροσώπηση σε διοικητικά συμβούλια και υπάρχουν και πολλές άλλες διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση ε, που συχνά δεν καταγγέλλεται ε, και δεν είναι μόνο θέμα ιδεολογία αυτό. Εδώ είναι θέμα βασική ανθρώπινη δικαιοσύνη. Πώ μπορούμε να ανεχτούμε μια τέτοια κατάσταση, όπου οι μισοί πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, δεν έχουν τι ίδιε ευκαιρίε για τη δουλειά του και για μια αξιοπρεπή ζωή. Ελπίζω λοιπόν η στρατηγική που προετοιμάζεται να μα επιτρέψει να ανταποκριθούμε σε αυτή την αυξανόμενη πίεση από το κοινό. Με κατάλληλα μέτρα. Πρόεδρος. Ο επόμενο ομιλητή, κυρία Γκάλβε Μουνιό, για ένα ε, λεπτό. Επίτροπε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία και που υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα όπως η διαφάνεια στους μισθούς, αλλά χαίρομαι κυρίως για το γεγονός ότι το θέμα του φύλου θα μπει στην Πράσινη Συμφωνία, στα θέματα της τεχνικής, της νοημοσύνης, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπήρχε πραγματικά συμπερίληψη τη διάσταση του φύλου στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Χρειαζόμαστε επίση πολιτική απασχολησιμότητα. Ε, θα πρέπει να εντάσσουμε δηλαδή του άνδρε και τι γυναίκε με τον ίδιο τρόπο στην αγορά εργασία, γιατί μέχρι στιγμή του εντάσσουμε με τελείω διαφορετικό τρόπο. Όσο δεν υπάρχει μια διάσταση του φύλου στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Επίση, αν δεν το καταφέρουμε στην οικονομική πολιτική, όπου λάμπει δια τη απουσία τη η διάσταση του φύλου δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή. Ούτε μία αναφορά. Επίτροπε Νταλή, ελπίζουμε να, υπάρξει, να δοθεί σημασία. Υπάρχει ένα δίκτυο για... με προσώπους ε, από όλες τις επιτροπές για το πώς θα λάβουμε υπόψη μας τη διάσταση του φίλου σε όλες τις πολιτικές, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μία πολύ πιο ίση Ευρώπη για όλους τους πολίτες της. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ε, η κυρία Μαξόβα, για ένα λεπτά. λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, στρατηγική της ισότητας των φύλων. Ε, είναι ένα πολύ δύσκολο φαρτό χαρτοφυλάκιο, αυτό το οποίο σας έχει ανατεθεί προκειμένου να προωθηθεί η στρατηγική αυτή. Θα πρέπει να ξεμπλοκάρουμε την, ε, ε, το ζήτημα της επικύρωσης στρατηγικής της, ε, της, Κωνσταντινού, της Συμφωνίας Κωνσταντινούπολης. Δυστυχώς η Τσεχοσλοβακία δήλωσε ότι θα αποσυρθεί. θα ήθελα να το ζητήσουμε ανοιχτά το θέμα αυτό και θα ήθελα να σας απευθύνω επίση μια έκκληση που σχετίζεται με το ζήτημα της εκπαίδευσης στα σχολεία. Η εκπαίδευση ξεκινάει πολύ νωρίς και είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό γιατί χωρίς αλλαγές στο σχολικό μας σύστημα, χωρίς ε, να... εάν δεν εξηγούμε στα παιδιά ότι η ισότητα είναι καθοριστική για την κοινωνία, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα. Έχουμε πάνω από 20 ε, συναδέλφους θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν είναι όμως, δεν είναι δυνατό να γίνει γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Παρακαλώ να επιδείξετε πειθαρχία. Θα είναι μόνο 4 αυτοί που θα πάρουν το λόγο. Ε, για ένα λεπτό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και ξεκινώ με τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Φίτζερ, στο πλαίσιο διαδικασία του Catch the Eye. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Επίτροπε Ντάλη, που ήρθατε να μας μιλήσετε για το μέλλον της στρατηγικής. Είναι πολύ σημαντική, είναι καλή η συγκυρία. Ε, έχουμε θετική επιτροπή. Δεν πιστεύω ότι μπορείτε μόνοι σας να κινηθείτε. Είναι σημαντικό κάθε επίτροπος να ασχοληθεί με το θέμα. Ε, πρέπει να ενσωματωθεί παντού η διάσταση του φύλου. Όλοι οι συνάδελφοι σκιαγράφησαν τα προβλήματα. Υπάρχουν και καινούργια θέματα, αλλά και παλιά που μας ταλαιπώρησαν καιρό. Πρέπει να προσέξουμε την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία την οικονομική κατάσταση των γυναικών. Πρέπει επίσης να δούμε και τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει ε, όλες οι αποφάσεις του προϋπολογισμού να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. Χρειάζονται και δεσμευτικά μέτρα και αυστηρή εφαρμογή όπως και παρακολούθηση και έλεγχος. Σας ευχαριστώ. Επόμενη. Μαρία Εμμανουέλα Μαρκές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη στρατηγική. Ελπίζω να περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα, στόχους και αντίστοιχους πόρους. Αλλιώς όλα αυτά θα μείνουν κενό γράμμα που θα μπει στα χρονοτούλαπα της Ένωσης. Χρειαζόμαστε στρατηγική για την καταπολέμηση των προβλημάτων, για να κερδίσουμε μάχες. Ε, υπάρχουν και ε, θέματα ενδοοικογενειακής βίας και αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε, να δούμε τι θα γίνεται στο μέλλον, αν η συμμεταχείριση ανδρών γυναικών στα τεχνολογικά επαγγέλματα. Υπάρχει μεγάλη ανισορροπία σήμερα. Όπως είπαμε, αυτή η στρατηγική θα πρέπει να ενταχθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής της Κομισιόν και οι επιχειρήσεις που έχουν καλά αποτελέσματα στον τομέα αυτό θα πρέπει και να ανταμείβονται. Ε, ελπίζω ότι αυτή η στρατηγική θα είναι φιλόδοξη και μπορείτε να υπολογίζετε σε μας και εμείς θα ταχθούμε στο πλευρό σας ενεργά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε η αξία που μπορεί να προσθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από τέσσερα στοιχεία. Το πρώτο, να υπάρξουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών και την καταπολέμηση της ανισότητας και, την βιότητα, και τη βία κατά των γυναικών. Δεύτερον, να βελτιωθούν οι στατιστικές και οι δείκτες προκειμένου να βελτιωθεί η αξιολόγηση αυτών των πολιτικών. Τρίτον, να θεωρήσουμε ότι η μάχη αυτή προποθέτει σφαιρικά κριτήρια αλλά και σε επίπεδο πολύ κοντά στο πολίτη, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε συνειδήσεις, να εφαρμόσουμε σφαιρικές ιδέες προκειμένου να αλλάξουν κάποια στερεότυπα που τροφοδοτούν ε, την ανισότητα στο επίπεδο του κάθε ατόμου. Ε, σημάδια ε, βίας ε, ενδοοικογενειακής, βίας κατά των γυναικών μόνο σε, μία χώρα μέλος θα έπρεπε να δώσουν λαβή στην ε, κατάρτιση μιας δήλωσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σίλβια Σαρδόνη έχει το λόγο. Μιλάμε εδώ για την ισότητα των φύλων. Στη χώρα μου, την Ιταλία, μόνο το 4% των διευθυντών είναι γυναίκες. Όμως το επίπεδο εκπαίδευσής τους είναι πολύ ψηλό παρόλα αυτά. Εδώ μιλήσαμε για μισθολογικές διαφορές. Είναι αναφίβολο, αλλά δεν νομίζω ότι η λύση είναι οι ποσοστώσεις. Δεν θέλω να με ορίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ε, δεν θέλω να γίνω ένα πάντα το οποίο θα προστατεύομαι μόνο και μόνο με γυναίκα. Θέλω να με αξιολογήσουν για τις ε, δυνατότητές μου, για τις δεξιότητές μου. Και αν είμαι καλύτερη από έναν άντρα, θέλω να πληρωθώ καλύτερα από τον άντρα, όχι το ίδιο με τον άντρα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να κλείσω την ομιλία μου λέγοντας ότι θέλω να αποφύγουμε αυτή την ε, συνεχή εκστρατεία των ανδρών υπέρ των γυναικών, να προβλέψουμε δηλαδή ποσοστώσεις ε, για να τις μεταχειριστούμε, λε και είναι κάτι το έθραστο, ένα μπιμπελό. Όχι, θα πρέπει να έχουμε γυναίκες να και να τους βλέπουμε ως άτομα, ως, ε, πολίτες και αν έχουν τις δυνατότητε να τις ε, επιβραβεύουμε γι' αυτό. Ο επόμενος ομιλητής, η κυρία Νόημαν. Κυρία Ντάλη, χαίρομαι πολύ που με τόση ενεργητικότητα μπαίνετε στο τομέα αυτό προκειμένου να χαραχθεί η στρατηγική αυτή, η οποία έχει και μια διάσταση εξωτερική πολιτική. Γιατί από τη μία η αλληλεγγύη μα ενισχύει, από την άλλη έχει αποδειχθεί ότι όσο περισσότερε γυναίκε ε, βρίσκονται στις εξωτερικές διαπραγματεύσεις τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Πολλές φορές μου είναι δυσάρεστο όταν πηγαίνουμε με την προσπίεση ε, του ΑΕΛΚ στο εξωτερικό και οι περισσότερες, ε, τα περισσότερα μέλη είναι άνδρες. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ εάν σε πλαίσιο αυτής της στρατηγικής δεν ε, ε, ασχολούνται μόνο στο επίπεδο της εσωτερική πολιτικής, αλλά ασχολούνται και με τις δικές μας τις δομές. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Η κυρία Τόμασίτς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. πολύ. Είναι σημαντική η ισότητα. Όλοι δηλαδή να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, να, κινούνται μέσα στο ίδιο σε ισότιμο πλαίσιο. Αλλά ίσες ευκαιρίες δεν σημαίνουν και ίση επιλογή. Η γυναίκα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τα ίδια επαγγέλματα με τους άνδρες και να έχει ίση αμοιβή, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό ε, θα το δεχτούν πολλές γυναίκες. Υπάρχουν και διαφορετικές αντιλήψεις ε, που έχουν να κάνουν και με τη, βιολογική ε, φύση της γυναίκας. Αν δημιουργούμε ίσες προϋποθέσεις δεν σημαίνει ότι θα αξιοποιηθούν αυτές. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορές, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Η μεταχείριση να είναι ίση. Αυτό είναι σαφές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ισότητα των γυναικών είναι, σημαίνει ότι θα ελέγχουν το σώμα τους οι γυναίκες. Εγώ χαιρετίζω την ε, πρόοδο στην Ιρλανδία, στην ε, Κύπρο, σε ό,τι αφορά την άμβλωση. Να προσέξουμε όμως, γιατί σε κάποιες χώρες έγινε προσπάθεια επιστοδρόμησης με αντιρρησίες συνειδήσεως που αντιμετωπίζονται άσχημα ε, και υπάρχουν πολλές φορές άδικες προϋποθέσεις, ακόμα και προσπάθειες απαγόρευσης της άμπλωσης. Προσοχή λοιπόν. Υπάρχουν γυναίκες μόνες που αντιμετωπίζουν πολλές διακρίσεις, οι Ρώμ, οι μετανάστριες. Ε, ε, αυτά θα πρέπει να τα αναδείξουμε, είναι σκάνδαλο. Στη Βουλγαρία έχουμε γυναίκες Ρωμά που είναι σε χωριστούς θαλάμους θα με ευτήρια. Δεν μπορούν να πάνε με άλλες γυναίκες. Θέλουμε συγκεκριμένες λύσεις γι' αυτό. Θέλουμε νομοθεσία η οποία θα απαγορεύει αυτές τις διακρίσεις και να βοηθήσουμε τις γυναίκες με κάθε δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λευτέρης Χριστοφόρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε οφείλω να πω ότι σε προηγούμενε ομιλίε μου η ευχή μου ήταν να μην χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε για θέματα ισότητα των δύο φύλων γιατί η ευρωπαϊκή ένωση θα μπορούσε να έρθει στο ύψο των περιστάσεων και αυτήν την ισότητα να την εφαρμόσει ίσα με σήμερα. θεωρώ προσβολή το ότι το 2020 η ευρωπαϊκή ένωση για την οποία περηφανευόμαστε για τον πολιτισμό τη για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τι αρχέ και τι αξίε και για κάτι που έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ισότητα των δύο φύλων συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε να το συζητάμε ω αν να είναι ένα στόχο ο οποίο οφείλουμε να επιδιώξουμε να τον κατακτήσουμε ενώ για τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να γίνει κάτι ορθωτό. άρα θεωρώ και πραγματικά επιβραβεύω την επίτροπο Ταλή για τι πρωτοβουλίε τη ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να μπει στην πρωτοπορία πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ούτω ώστε να επιβληθεί αυτή η ισότητα στι χώρε εκείνε που δεν τον εφαρμόζουν με κυρώσει να υπάρξει ακόμα και στήριξη αυτή τη προσπάθεια και μέσα από του προπολογισμού και να βγει αν είναι δυνατόν μια οδηγία από την ευρωπαϊκή ένωση ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο ισότητα των δύο φύλων η ευρώπη τελειώνοντας ευρώπη και μη εξάλληψη της διάκρισης της βίας κατά των γυναικών δεν νοείται και δεν μπορεί να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. άρα είναι πρώτος και μοναδικός στόχος να το πολεμήσουμε μαζί. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Χάιζελ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να βασίζεται σε αυτές τις αξίες και να είναι μεγάλη έμπνευση για τις μελλοντικέ γενιές. Θα πρέπει να είναι πολιτική δέσμευση για τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να έχει και κάποια στοιχεία πολιτικών δεσμεύσεων. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι αδιανόητο οι γυναίκε να πληρώνονται λιγότερο από του άντρε. Επίση, στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να έχουμε γυναίκε που παίρνουν λιγότερα, που παίρνουν λιγότερα λεφτά τους άντρες. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες να βρίσκουν θέσεις στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τους. Θα πρέπει να είναι εύκολη πρόσβαση και να είναι και φθηνή. Ε, επίσης πρόσβαση στο, στην περίθαλψη, υγειονομική περίθαλψη. Θα πρέπει να λυθεί αυτή η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές βίας, σεξουαλικής, ενδοοικογενειακής, στην εργασία. Ε, θα πρέπει να πολεμήσουμε ακόμα και τα δυσάρεστα σχόλια κατά των γυναικών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρτιτς είναι ο τελευταίος ομιλητής. Έχει ένα λεπτό. Η διάκριση των ε, περισσότερων ε, γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, την απασχόληση και την επαγγελματική σφαίρα μέχρι τον ιδιωτικό βίο. Είναι απαράδεκτη και δεν συνάδει με τις ε, θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Νομίζω ότι δεν δείχνουμε αρκετή αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Η... Χθες ήταν η Διεθνής ημέρα των γυναικών. Φοβούμαι ότι ακόμα και στο κοινοβούλιο αυτό οι περισσότεροι περιορίζονται σε ρητορικά σχήματα. Ε, βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι ε, του ΕΛΚ ε, απορρίπτουν, καταψηφίζουν σημαντικά και ε, τροπολογίες ε, που τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε καταπηγόντως διαφορετικά μέτρα. Χωρίς μια μελλοντική στρατηγική για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, ε, θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε κενές εξαγγελίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. μία χώρα η χώρα, στη χώρα μου οι γυναίκες ζουν σε πολλές περιοχές της υπαίθρου. Ε, ε, μόνο 1% των, γυναικ... των ανδρών παίρνουν πατρική άδεια. Ε, μιλάω για την Πολωνία. Δεν υπάρχει το δικαίωμα στην έκτρωση. Η... Ε, και η κατάσταση επηρεάζει περισσότερο αρνητικά γυναίκες με αναπηρία ή την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ τον 21ο αιώνα στο κέντρο της Ευρώπης είναι απαράδεκτο να υπάρχουν γυναίκες που δεν μπορούν να έχουν τα εξασφαλισμένα τα απολύτως θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ενοποιημένες προδιαγραφές και υψηλό επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες μέλη. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας στόχος της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων. Ευχαριστώ. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επίτροπος Ντάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις σημαντικές συνεισφορές σας. Ναι, είμαστε στο 2020 και ακόμα συζητάμε τα δικαιώματα του 50% και πλέον του παγκόσμιου πληθυσμού. Συζητούμε τα δικαιώματα που οι άντρες τα θεωρούν δεδομένα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πραγματικά όλους για τις εκκλήσεις και τη διάθεση περισσότερων ανδρών να συμμετάσχουν στη συζήτηση για την ισότητα των φύλων. Όλοι έχουμε μητέρες, μερικοί από εμά έχουν κόρες και εκφράζουμε το 50% και πλέον του πληθυσμού και το εκπροσωπούμε. Ένας άντρας μάλιστα είπε ότι ο φεμινισμός δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, είναι υπόθεση ολόκληρης κοινωνίας. Επομένως, βεβαίως, ο κύριος Μπιεντρών πολύ σωστά το είπε, ότι όταν συζητάμε τους εξοπλισμούς και τον πόλεμο, που σκοτώνουν ανθρώπους όπως εσείς και εγώ, οι περισσότεροι που ομιλητές είναι άντρες. Δεν θέλω περισσότερες γυναίκες να συνεισφέρουν σε τέτοιου τους συζητήσει. Αλλά τουλάχιστον έχουμε λιγότερους άντρες που μιλάνε για αυτά τα θέματα. Και θέλω όλοι μας, όλοι μαζί, να συζητούμε την ειρήνη. Αλλά δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό και να ασχοληθούμε με την ισότητα των φύλων και να θεωρήσουμε ότι μας αφορά όλους, όλες τις κοινωνίες μας, όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο. Η νέα στρατηγική για την ισότητα των φίλων θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα σημεία, όλα αυτά τα θέματα που τονίσατε και αυτό που αναφέρουν οι πολιτικέ κατευθύνσει τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε μια φιλόδοξη ατζέντα, ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την καταπολέμηση όλων των μορφών βία ε, και την βία στο διαδίκτυο. Θα παρουσιάσω μια νομοθετική πρόταση, ούτω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για του μισθού στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, και θα λάβω και άλλα μη νομοθετικά μέτρα για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών. Θέλω ευρωπαϊκού κανόνε, ούτω ώστε να υπάρχει πρόοδο στην ισορροπία ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Γιατί ξέρουμε ότι οι στόχοι δίνουν αποτελέσματα. Θέλω η οδηγία για τη συμφιλίωση οικογενειακή και επαγγελματική ζωή να πρέπει να εφαρμοστεί, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη, να πούμε, και του άντρε και τι γυναίκε και να συμφιλιώσουν τι ζωέ του. Θέλω όλε τι πρωτοβουλίε να αξιολογούνται επίση και από τη σκοπιά τη ισότητα των φύλων. Η δουλειά της Κομισιόν για την ε, ένταξη της διάστασης του φύλου στι πολιτικέ θα να, είναι πιο, να γίνεται πιο συστηματικά, να αγγίζει περισσότερα θέματα από ό,τι συνέβαινε μέχρι τούδε. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στη διάσταση του φύλου όταν μιλάμε για βασικά προβλήματα της ε, κοινωνίας ή θέματα της κοινωνίας και προκλήσεις, όπως ψηφιοποίηση και μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Το ανέφεραν και κάποιοι ευρωβουλευτές. Και ναι, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι οι, περισσότερες οι περισσότεροι φτωχοί είναι γυναίκες. Και είναι συχνά αποτέλεσμα ε, πολλών ανισοτήτων, σειρά και σωρία ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν κορίτσια και γυναίκε καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Βασίζομαι στην ισχυρή στήριξη του Κοινοβουλίου, γιατί η ισότητα για όλου του πολίτε είναι μία από τις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να την υλοποιήσουμε αυτή την αξία όλοι μας για όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Κλείνει αυτή η συζήτηση. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης. Προφορική ερώτηση για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 64η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας. Να σας υπενθυμίσω ότι για να πάρετε το λόγο να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παραδοσιακό ή το ηλεκτρονικό σύστημα. Οι οδηγίες υπάρχουν στην είσοδο της Αυσίας Ολομέλειας. Και τώρα το λόγο έχει στην ε, πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, την κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, γιορτάζομαι την 64η επέτειο ενός κειμένου ε, πρωτόγνωρου. Η δήλωση του Πεκίνου που εγκρίθηκε στη διάσκεψη εκεί είναι από τα πιο προοδευτικά έγγραφα για τα δικαιώματα των γυναικών. Όλοι οι τομείς της ζωής καλύπτονται. Πλήρης ισοτιμία ε, είναι ο στόχος. Ε, είτε πρόκειται για πλούσιες γυναίκες, είτε γυναίκες που ζουν σε μπόλεμες ζώνες ή σε ειρηνικές. Ε, το 1995 όλοι αναγνώρισαν τα δικαιώματα της γυναίκας ως ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν μια μάγνα κάρτα των γυναικών που θέτει τις γυναίκες στο, σε ίση με τους άνδρες. Ε, όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις συμβάλλουν για την υλοποίηση της διακήρυξης. Ε, ε κυβερνήσεις τάχθηκαν ε, και δεσμεύτηκαν υπέρ της ε, των δικαιωμάτων των γυναικών και προβλέπουν τακτικούς ελέγχους της κατάστασης. Επίσης, η, ισότητα των γυναικών σε θέσεις ε, εξουσίας, η ε, και αυτό συμπεριλαμβάνεται. Επίσης, ε, βασική ε, προϋπόθεση για την ισότητα είναι να έχει την εξουσία η γυναίκα όχι μόνο στην επαγγελματική ζωή, αλλά και στην δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις για τον εαυτό της. 25 χρόνια μετά από την ε, διακήρυξη ε, τα αποτελέσματα δεν είναι ε, τόσο ενθαρρυντικά. Η αυτοδιάτηση των γυναικών δεν είναι κατοχυρωμένη ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς διαπιστώνουμε ότι χρειάζονται ε, μέτρα για την ε, ίση θέση των γυναικών. Δεν ε, μπορούμε να περηφανευόμαστε θα πρέπει να προωθήσουμε ένα θέμα που έχει μπλοκαριστεί επί 8 χρόνια, δηλαδή έλλειψη εκπροσώπησης, διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Δεν υπάρχει πρόσβαση στα ε, ε, ισότιμες στις υπηρεσίες ε, επίσης, οι αμοιβέ. Βλέπουμε ε, ότι οι καθαρές αμοιβέ ε, αποκλίνουν ακόμα πολύ. 500.000, μισό εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια πέφτουν θύματα κροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Και αυτά και μέσα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι συντριπτικά στοιχεία το Συμβούλιο, οι, οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένα να βοηθήσουν το μισό του πληθυσμού, ε, να του στηρίξουν, ούτως ώστε να επιτευχθεί πλήρης ισότητα. Ε, τα παραδοσιακά, θρησκευτικά και άλλα στερεότυπα ε, ε, παρεμποδίζουν την επίτευξη της ισότητας και οι πατριαρχικές δομές δεν αφήνουν τη γυναίκα να γίνει ισότιμη. Πρέπει να δοθεί μάχη λοιπόν σε αυτό. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε με κανένα τρόπο οπισθοδρόμηση στην κατάσταση που έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί. Προειδοποιώ, πρόκειται για το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ε, που δεν έχει ε, ε, κατοχυρωμένα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι γυναίκες τώρα έχουν ένα έγγραφο στα χέρια τους που διασφαλίζει τη διεθνή νομιμότητα. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει τώρα να πάρει πνοή. Τα, ε, ε όλα τα έθνη θα πρέπει να ε, συνεργαστούν ε, για μία πλήρη υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται. Χρειάζεται πρακτική εφαρμογή. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στους αγαπητούς συναδέλφους να ε, ψηφίσουν ε, υπέρ των προτάσεων που κάνω. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε ισχυρή συμμετοχή και πολύπλευρη προσέγγιση. Τα Ηνωμένα Έθνη ζουν από τη συνεργασία, την κοινή βούληση και την κοινή δράση. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και εμείς να παρουσιαστούμε ενωμένοι στη διαφορετικότητά μας. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Νικολίνα Μπρντάτς, παρακαλώ, για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία να αλλάξουμε τις απόψεις, να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά την 64η Σύνοδο της Επιτροπής του ΙΕ, τη θέση της γυναίκας. Ε, το 2030 είναι το έτος για την υλοποίηση της ισότητας των φύλων και, ε, το 2020, συγγνώμη, και θα είναι ένα ορόσημο όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Ε, θα εορτάσουμε την επέτειο της, της, ε, την 64η Σύνοδο της Επιτροπής ε, του ΟΗΕ και την 25η επέτειο της δήλωσης του Πεκίνου. Ζητήματα ισότητας φύλων αφορούν όλους τους πολίτες, όχι μόνο θέματα των γυναικών. Πρόκειται για ένα κοινωνικό και οικονομικό θέμα που επιτρέπει σε όλους ίσες ευκαιρίες προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη σημαντικών ωφελιών και, ενίσχυση, και ε, οικονομική ενίσχυση. Στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής πει σε σχέση με το στάτους των γυναικών θα πρέπει να επισημάνουμε τις ελλείψεις όσον αφορά την υλοποίηση της ε, συμφωνίας του Πεκίνου και θα πρέπει να επικυρώσουμε το βαθμό ε, υλοποίησης ε, των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει εδώ και πέντε χρόνια. θα πρέπει οι γυναίκες να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα η πρόοδος ε, σε πολλούς ε, τομείς, όπως ελέγχθη, ε, στερεί. Πολλές γυναίκες εκτίθενται σε ακραία φαινόμενα βίας και φτώχειας. Ε, παραμένει μισθολογικό χάσμα σε εργασιακό επίπεδο και υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών σε, σε ηγετικές θέσεις σε όλους τους τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση στερεί ως προς όλους αυτούς ε, τους τομείς. Αυτό θα πρέπει να εξισορροπηθεί. Ε, όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις για την πολιτική δήλωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατράνωσε την αποφασιστικότητά της για να πετύχει ισότητα των θέσεων και κάτι το οποίο δράζεται στο νομικό πλαίσιο της Ευρώπης. Ορισμένα από τα πιο κρίσιμα θέματα περιλαμβάνουν τα εξή. Ισότητα και μη απάλληψη των διακρίσεων, ε, βία κατά των γυναικών, ε, πολιτικές προσαρμοσμένε προς την οικογένεια, ε, κοινωνική προστασία, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι η βάση της, της νέα προσέγγιση. Θα πρέπει επίση να υπάρξουν κατευθυντήριε γραμμέ ε, για την κλιματική αλλαγή και τι ε, τεχνολογίε επικοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κατοχυρώσει τα υπάρχοντα επιτεύγματα και να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Επίσης ε, προσπαθεί μια, να κάνει μια πολιτική δήλωση η οποία ε, κατοχυρώνει επίσης τους ακτιβιστές υπέρ των ε, δικαιωμάτων των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται μια πλήρη υποστήριξη προς τις ΜΚΟ ε, προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε τοπικό, εθνικό και σφαιρικό επίπεδο. Όσον αφορά τι πολιτικέ δηλώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανακτήρια συνεδρία, είμαστε πεπισμένοι ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, μοιράζονται τι ίδιε προτεραιότητε και τι ίδιε αξίε. και περιμένουμε με ανυπομονησία τι δικέ σα προτάσει και υποδείξει. Ε, Αξιότιμα μέλη, όσον αφορά ευρύτερα το ζήτημα της ότητας των φύλων, τονίσατε το γεγονός ότι η πολιτική φύλου δεν είναι μια διακριτή, ένας διακριτός πολιτικός τομέας, αλλά αφορά όλες τις, όλους τους ε, τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτοχρόνως, άπτεται όλων των σημαντικών ε, στρατηγικών. Χρειαζόμαστε μια συμπερίληψη διάσταση στους φίλους σε όλους τους πολιτικούς τομείς. Στα συμπεράσματα του περασμένου Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια στρατηγική υψηλού επίπεδου για την ισότητα των δύο φίλων Και χαίρομαι που ανέλαβε η Επιτροπή το έργο αυτό. Το Συμβούλιο ε, ε, ε, σας καλεί να μεριμνήσετε για ε, μια συμπερίληψη της διάστασης του φίλου σε όλους τους τομείς ε, και καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει την προσοχή της περισσότερο στην ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τέλος, ορισμένα πράγματα σε σχέση με το έργο του Συμβουλίου ε, χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες που εξήγηλε η Επιτροπή όπως μέτρα που βασίζονται στην διαφάνεια όσον αφορά τις ε, πληρωμές, τις αμοιβέ. Ε, καταπολέμηση των διακρίσεων είναι μία από τις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας. Θέλουμε να υποβάλουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, προκειμένου να πετύχουμε μία ισορροπία. Ε, οι γυναίκες... Ε, έχουν περιορισμένες δυνατότητες συμμετοχής ε, στην αγορά της εργασίας. Ε, στις 4 Δεκεμβρίου, στις 30 Ιανουαρίου θα διοργανώσει μια συνδιάσκεψη που τα αποτελέσματά της θα συζητηθούν με την Επιτροπή των Γυναικών γιατί πολλά πράγματα έχουν γίνει παρόλα αυτά υπάρχει μπροστά μας μακρύς δρόμος προκειμένου να εξασφαλίσουμε πλήρη ισότητα ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πέρα από τα όρια της. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επίτροπος Ντάλη. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι βουλευτέ. Σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε την προετοιμασία της 64ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Είναι τέλειος ο χρονισμός. Οι διαπραγματεύσεις για την πολιτική δήλωση και την προετοιμασία της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι εν εξελίξη. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει η σύνοδος με μία ισχυρή πολιτική δήλωση που να μιλάει για τις δράσεις που πρέπει να αναλυθούν και να μιλάει για την εφαρμογή των ε, δεσμεύσεων που έχουν αναλυθεί. Παράλληλα, ε, ετοιμάζουμε και διάφορες εκδηλώσεις που θα είναι ένα χωνευτήρι καλών πρακτικών, νέων ιδεών για το πώς το θεματολόγιο του Πεκίνου θα προχωρήσει, θα εφαρμοστεί. Αυτή είναι η δύναμη Τη συνάντηση αυτή, τη συνόδου αυτή. Συναντόμαστε με πολλούς εταίρους και συζητάμε για την ισότητα των φύλων. Στη σύνοδο αυτή γιορτάζουμε την 25η επέτειο της δήλωσης του Πεκίνου και της πλατφόρμας για δράσεις. Επίσης χαιρόμαστε την 25η ε, σύνοδο του ΟΗΕ και την 5η σύνοδο για τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Η ισότητα των φίλων, η ενίσχυση των γυναικών και των κοριτσιών δεν είναι θέμα μόνο δικαιοσύνη. Έχει οικονομική έννοια να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρε, τα κορίτσια και τα αγόρια, υλοποιούν το δυναμικό που έχουν. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση της ε, Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ για την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών παντού στον κόσμο. Είναι μια έκθεση με πολλές αποχρώσεις. Ε, έχουν ε, εξεταστεί οι εθνικές καταστάσεις 167 ε, χωρών και έχουν γίνει πολλές συνεδριάσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη για να ετοιμαστεί αυτή η έκθεση. Και ενώ υπάρχει πρόοδος, δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε. Η αγορά εργασίας των γυναικών, μάλλον η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί, αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια έχει βαλτώσει οι γυναίκε έχουν υπερβολικέ φροντίδε ε, στο σπίτι. Ε, η φωνή των γυναικών και των κοριτσιών δεν ακούγεται τόσο χειρά όσο των ανδρών και αγοριών. Οι γυναίκες είναι 25% πιο πιθανό να ζουν σε συνθήκες στόχια στη ζωή τους. Τα στερεότυπα του φίλου καθορίζουν τι κάνουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στη ζωή τους. Ε, η βία εναντίον κορισιών και γυναικών είναι ένα θέμα που βλέπουμε ξανά και ξανά. Επίση, έχουμε παράλληλα τώρα τι ψηφιακέ τεχνολογίε, διάφορε αλλαγέ. Αυτέ οι αλλαγέ θα πρέπει να γίνουν ευκαιρία. Η ψηφιοποίηση μπορεί να ανοίξει πόρτε για τι γυναίκε και τα κορίτσια, αλλά μπορεί επίση να χρησιμοποιηθεί λάθο για να τι φημώσει. Όπω είπε ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών είναι σημαντική για έναν οικονομικά σίγουρο κόσμο όπου η πόλωση αυξάνεται και οι περιβαλλοντικές ε, συγκρούσεις και απειλές αυξάνονται επίσης. Η ο άνισος καταμερισμός της εξουσίας διαιωνίζουν τις ανισότητες του φύλου. Καλωσορίζω την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και το ψήφισμά σας που θα δημοσιευθεί ως Νούπο για αυτό το θέμα και την παρουσία του ε, Κοινοβουλίου στην εκδήλωση αυτή ε, του ΟΗΕ. Είναι προτεραιότητα αυτή ισότητα των φύλων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσωτερικά, αλλά και στις εξωτερικές μας σχέσεις και δράσεις. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων τον Μάρτιο και το 2020 θα ετοιμάσει το τρίτο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις. Μια φιλόδοξη, ισχυρή προσέγγιση που θα αντιμετωπίζει τα παγκόσμια προβλήματα και τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βασιστούμε στην ένταξη του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Η Task Force για τις ανισότητες με μέλη από όλες τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα είναι σημαντική και θα κάνει σημαντική δουλειά. Επίσης, στοχευμένες δράσεις για συγκεκριμένα θέματα ισότητας των φύλων θα συνεχιστούν. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε το μισθολογικό χάσμα και θα υπάρχει διαφάνεια για τους μισθούς. Μισθούς και θα αναπτύξουμε μέτρα για να σταματήσουν ε, οι ανισότητες στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Προσβλέπω σε γόνιμη συζήτηση. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις ιδέες και σας ευχαριστώ που βάλατε τη συζήτηση αυτή στη σημερινή μερίσια διάταξη. Ευχαριστώ. Επίτροπε, και τώρα από το ΕΛΚ η κυρία Francis Fitzgerald. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω τις δύο ομιλίες, τρεις ε, και της Εύελιν σκιαγραφούν σαφώς τις προτεραιότητες που πρέπει να παρουσιάσουμε στη διάσκεψη του ΟΗΕ. Η γλώσσα είναι σωστή, οι λέξεις σωστές και μπορούμε να προωθήσουμε τις προτεραιότητες που έχουμε προδιαγράψει, προτεραιότητες ε, που πρέπει να υποβάλλουμε στον ΟΗΕ. Πρόοδος έχει επιτελεστεί αλλά υπάρχουν ακόμα πολύ σοβαρά θέματα που πλήττουν τις γυναίκες. Σημειώνουμε ότι μετά τη διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη, οι δεν υπέγραψαν στο τέλος τη δήλωση, στο τέλος της διάσκεψης και αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Τώρα έχουμε ε, την 25η ε, επέτειο ε, που για τα δικαιώματα των γυναικών της Χίλαρη Κλίντον πρόκειται για επιτάχυνση, εφαρμογή, στόχους και παρακολούθηση. Επίσης πρόκειται και για τον προϋπολογισμό. Είναι σημαντικό το στοιχείο αυτό για τις συζητήσεις φέτος στον ΟΗΕ. Επίσης ε, πρέπει να προσέξουμε ε, στάσεις ε, κυρίαρχες πολλές φορές, καθημερινού σεξισμού και αυτό πρέπει να το δούμε. Αντίληψη για τις γυναίκες, οι ε, αναφορές για τις γυναίκες και ακούσαμε και επικρίσεις ε, ε, για τις ποσοστώσεις τι λέει ο ΙΕ, ότι είναι προσωρινό αναγκαίο μέτρο. Οι ποσοστώσεις λειτουργήσαν για πολύ καιρό υπέρ των ανδρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Φριτσόν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε όταν είχα πάει τελευταία στη Νέα Υόρκη, στην Επιτροπή για τις Γυναίκες του ΟΗΕ, και ε, ήταν ντροπή που δεν είχε στρατηγική για την ισότητα η Ένωση. Τώρα θα εκπροσωπήσω με το Κοινοβούλιο και θα φροντίσουμε η Ένωση να πάρει το θέμα στα σοβαρά τώρα με την στρατηγική της Επιτρόπου Ντάλι. Οι γυναίκες ε, συνέρχονται στον ΟΗΕ, αυτό είναι σημαντικό. Οι γυναίκες ε, συμβάλλουν στις ε, ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και ήδη χαίρομαι που θα συμμετάσχω στην Επιτροπή των Γυναικών. Είναι σημαντικό να ζητήσουμε ε, τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Χρειαζόμαστε και προοπτική ίσης ε, ισότητας και στον τομέα του κλίματος. Αυτό είναι σημαντικό και για τις γυναίκες, για τα παιδιά, για τα κορίτσια και για τους άνδρες όμως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, για την ομάδα Αρινιού, η κυρία Σεμίρα Ραφαέλα, δύο λεπτά. Κυρία Επίτροπε, τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Ζούμε, ε, δεν πρέπει να ζούμε σε έναν κόσμο που πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Οι άνδρες και οι γυναίκες της παλιάς και της τωρινής γενιάς δούλεψαν σκληρά για να φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο σε αυτά τα θέματα. Δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα αυτά τα δικαιώματα. Και την δημοκρατική μας κοινωνία στην Ευρώπη δεν πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη. Υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις. Υπάρχουν ε, οργανωμένα συμφέροντα κατά των γυναικών. Εμείς πρέπει να αναδείξουμε τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει και να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας για μια πιο κοινωνική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες και οι γυναίκες. Αυτή η πρόταση ψηφίσματος είναι η δική μας δέσμευση ε, στην ε, σύνοδο του ΟΗΕ για την ενίσχυση των γυναικών. Είναι σημαντικό το όραμα. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να θέσουμε στην πράξη τις δεσμεύσεις μας ε, για την Ατζέντα 2030. Η ισότητα είναι σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2020 είναι το έτος της ε, εφαρμογής της ισότητας και της ενίσχυσης γυναικών και κοριτσιών. Εγώ χαιρετίζω τη στρατηγική της ε, ε, Επιτρόπου Ντάλη. Στο τέλος Μαρτίου γιορτάζομαι την επέτειο των κατοχήρωση δικαιωμάτων των γυναικών. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε τη μάχη για βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών και της θέσης, στην, θέση, στον χώρο της εργασίας. Η Κομισιόν πρέπει να κάνει τα πάντα ούτω ώστε οι γυναίκε να αναδείξουν όλο το δυναμικό τους, να έχουν πλήρη πρόσβαση στην εργασία και ίσες ευκαιρίες που παρέχει η κοινωνία μας. Α συνεχίσουμε να ε, δίνουμε μάχη γι' αυτό και να ακούμε τη φωνή των γυναικών παντού ε, η συμμετοχή μας στην, 20, στην 64η Σύνοδο δείχνει ότι όλα αυτά τα παίρνουμε πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα για την ομάδα ID η Κριστίνα Άντερσον για 1,5 λεπτό. Το Κοινοβούλιο ε, ε, μιλάει τώρα για τη θέση που θα λάβει στην 64η Σύνοδο. Τα δικαιώματα των γυναικών μπορούν να ενισχυθούν μόνο αν θεωρηθούν ε, ως ε, μέσω τη εκ των υστέρων. Ε, ε, τα δικαιώματα των, της κοινότητας των ΛΟΑΔ πρέπει να είναι κατοχυρωμένα και οι γυναίκες προβλέπεται ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε ποσοστώσεις για να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε, ε, ε πώς είναι δυνατόν όμως, τι σεξιστική αντίληψη είναι αυτή ότι οι γυναίκες δεν μπορεί να προωθηθούν χωρίς την, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να φροντίσουμε ε, να καταλάβουμε ότι οι γυναίκες ε, δεν τα χρειάζονται όλα αυτά. Ε, είναι πολύ σημαντικό να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα στον ε, δημόσιο χώρο. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για διαφορετικότητα, για ανεκτικότητα ε, όταν παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Ως γυναίκα στην Ευρώπη έχω ελεύθερη διακίνηση, όπως και οι άνδρες. Πριν λοιπόν μιλήσουμε για γελίες ποσοστώσεις στα ψηφίσματά μας, και ε, ασχολούμεθα με αυτά όλα τα δευτερεύοντα, αναρωτιέμαι εδώ ε, πώς, ε, τι κάνουμε στο Κοινοβούλιο για να προστατέψουμε αυτούς, ε, αυτές που ζητούν προστασία όντως. Η επόμενη ομιλήτρια η κυρία Βάνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό που δείχνει η συζήτηση είναι αυτό που μας ενώνει ως Κοινοβούλιο, Κομισιόν και Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε στον ΟΗΕ με ενιαία φωνή ε, και να αντιπαρατεθούμε ενάντια στις προσπάθειες οπισθοδρόμησης. Να δώσουμε μάχη για διεθνή ισότητα σε όλους τους τομείς για τις ε, γυναίκες. Η διακήρυξη του Πεκίνου είναι το ευρύτερο φόρουμ ε, για να κινηθούμε. Εμείς ως Ευρωπαίες έχουμε την υποχρέωση να ε, τεθούμε στο προσκήνιο των πολυμερών δράσεων. Εμείς οι, Ευρω... οι γυναίκες και ε, εμείς οι Ευρωβουλευτές ε, αύριο θα εγκρίνουμε ένα ψήφισμα σχετικό και ελπίζω ότι και το Συμβούλιο που καλείται ε, να λάβει σαφή θέση επίσης να το κάνει και να προσχωρήσει την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και να πάρει σαφή θέση για την ισότητα των φίλων. Ευχαριστώ. Κυρία Βυσνιεύσκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και τη σότα των Φύλων ε, κάνει διακρίσεις εναντίον των μικρών πολιτικών ομάδων. Στην ετήσια σύνοδο που γίνεται στην Νέα Υόρκη. Είσαστε ικανοποιημένοι με κάτι τέτοιο η φωνή των συντηρητικών γυναικών σε αυτή τη διάσκεψη δεν θα ακουστεί. Αυτέ που θέλουν να συνδυάσουν την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Αυτοί που δεν θεωρούν ότι το γάμο και η μητρότητα είναι βάρο που θα εμποδίσει τι καριέρε του. Η φωνή που λέει ότι η ζωή είναι ένα θαύμα και πρέπει να προστατευτεί. Ε, αυτή η φωνή δεν θα ακουστεί. Όμω η ζωή έχει ψηλή αξία. Μόνο οι αριστερέ και οι φιλελεύθερε φωνέ θα ακουστούν η χειρά. Αυτές που λένε ότι η άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ότι είναι ένας τρόπος για να κάνεις οικογενειακό προγραμματισμό. Ε, οι, φωνές, που χειραγωγούν ε, τις απόψεις και τα θέματα του φίλου. Με αυτές τις ιδεολογίες δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Ψηφίστε το ψήφισμα, σας παρακαλώ, του ECR. Η κυρία Ροντρίγκε Πάρλο. Κυρίες και κύριοι, παρουσιάζουμε μια πρόταση ψηφίσματος όπου υποβάλλουμε μια σειρά συστάσεων που θεωρούμε ότι έχουν προτεραιότητα όσον αφορά τη θέση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, στο βέβαιο είναι ότι μέχρι στιγμή δεν σα έχει κινητοποιήσει ιδιαίτερο στο ζήτημα του φεμινισμού. Το ε, Συμβούλιο είναι το όργανο το οποίο μπλοκάρει την πιο σημαντική πρωτοβουλία για τι γυναίκε. Για παράδειγμα, μια οδηγία κατά των διακρίσεων που έχει μπλοκαριστεί εδώ και 10 χρόνια στο Συμβούλιο. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι ε, ο βηματισμό είναι αυτός τη χελώνα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επικυρώσει το, τη δήλωση της Κωνσταντινούπολης λόγω της πίεσης που ασκεί η ομάδα χωρών του Βίζεκρατ, η η θρησκευτική κύκλη ε, σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Ε, οι γυναίκες θεωρούνται ως αναπαραγωγικές ε, μηχανές ε, στην υπηρεσία των ανδρών ή των κυβερνήσεών τους. το Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι μία αναγνώριση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας δεν είναι μία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και αυτό συνάδει με την θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εγκρίνει μια οδηγία σε σχέση με την ε, βία ε, του φίλου. Το Κοινοβούλιο έχει ε, αναγνωρίσει